Ε, είμαι ευγνώμων στου συναδέλφου που μίλησαν και θα μεταβιβάσω το μήνυμά σα στους άλλου εταίρου στην ε, G20. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα σα ευχαριστώ Επίτροπη κυρία Άντορ. Εδώ ολοκληρώνω τη συζήτηση του θέματο. Το επόμενο σημείο της σημερινής είναι η δήλωση τη Κομισιόν για την καταπολέμηση τη φυματίωση. Μπορούμε να χαιρετήσουμε τον Επίτροπο Ντάλι και να του δώσουμε το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, εξότιμοι ευρωβουλευτές, χαίρομαι που μου δίνετε την ευκαιρία αυτή να έρθω εδώ σήμερα για να υπογραμμίσω την δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις από την ασθένεια αυτή, τη φυματίωση. Εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχουν ακόμα απειλές από την ασθένεια αυτή για τη δημόσια υγεία. Είχαμε πιστέψει ότι είχαμε επιτυχίες, αλλά το πιστέψαμε αυτό για πολύ καιρό. Κάναμε λάθο όμω και δεν προστατευτήκαμε αρκετά από τη φυματίωση. Το 2008 το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Πρόληψη Ασθενειών και τον έλεγχο των ασθενειών ανέφερε 83.000 περιπτώσει φυματίωσης και 6.000 θανάτου εξαιτία τη ασθένεια αυτή τη φυματίωσης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι χώρε Εζέ. 16 θάνατοι τη μέρα. Είναι απαράδεκτο και απαιτεί δράση από όλες τις πλευρές είναι απαράδεκτο γιατί η φυματίωση είναι μια ασθένεια που θεραπεύεται και που προλαμβάνεται και που δεν πρέπει να οδηγεί σε τέτοιες τραγικές συνέπειες. Η φυματίωση συνδέεται με πολλές από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα. Δεν έχουμε νέα μέσα για την διάγνωση και την έγκαιρη είναι μεταδοτική και σίγουρα πλήττει δυσανάλογα πολύ τους ε, λιγότερο εύπορους. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες που έχουν αναλυθεί τα τελευταία χρόνια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την φυματίωση. Το 2000 η φυματίωση συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο των ασθενειών κατά προτεραιότητα και στα πλαίσια αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριξε πολλά προγράμματα τα οποία φρόντιζαν για το συντονισμό των δράσεων κατά της φυματίωσης ε, στις ε, χώρες ε, που έχει ορίσει Διεθνής ε, Οργάνωση Υγείας, Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Μέσω των ερευνών επίσης που γίνονται, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει την ανάπτυξη εμβολίων, νέων μέσων θεραπείας, διαγνωστικών μέσων επίσης για τη θυματίωση. Από το 2002 και μετά έχουμε δώσει πάνω από 24 εκατομμύρια για το λόγο αυτό. Η θυματίωση όμως δεν έχει σύνορα. Γι' αυτό και πρέπει να στηρίξουμε χώρε πέρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει αναπτυσσόμενε χώρε για να καταπολεμήσουν την φυματίωση μέσω προγράμματο για να αντιμετωπιστεί η ασθένεια αυτή, όπω επίση και η ελαιονοσία. Τα κύρια κανάλια για να αντιμετωπιστεί το AIDS, η φυματίωση και η ελαιονοσία με 170 εκατομμύρια από το 2002 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προσπαθεί να στηρίξει τα προγράμματα αυτά. Επίσης ε, στηρίζει και άλλα προγράμματα στην Αφρική και άλλες ε, αναπτυσσόμενες χώρες. Τέλος, η δημιουργία Ευρωπαϊκού Κέντρου για την πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών μας επιτρέπει να κάνουμε περισσότερε προσπάθειε ακόμα για να απαλληφθεί η φυματίωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από έτοιμα της ε, Κομισιόν, το Κέντρο Πρόληψης έχει αναλάβει νέα μέτρα με, αντιμετωπίζοντας πολλαπλές προκλήσεις που οδηγούν στην ε, φυματίωση ενισχύοντας τους ελέγχους. Επίσης θέλουμε φροντίδα για όλους, νέα μέσα για τη διάγνωση και την θεραπεία, μείωση του βάρους από την μετάδοση της φυματίωσης ε, και του AIDS, αλλά η Επιτροπή δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνη της τις προκλήσεις αυτές. Χρειάζεται η βοήθεια της κοινωνίας των πολιτών, ε, προστατεύοντας τους πιο ευάλωτους. Τα κράτη-μέλη επίσης παίζουν ρόλο κλειδί προκειμένου να καταπολεμηθεί η ασθένεια αυτή. Ευχαριστώ κύριε Πέτρο Καταλή. Εξ νόμου των πολιτικών ομάδων έχουμε τους ομιλητές τώρα. Καταρχήν η κυρία Αντωνέσκου για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε. Την εποχή των αντιβιωτικών είναι αίτιο θανάτου. Έτσι χαρακτήρισαν την φυματίωση κάποιοι ειδικοί. Ήταν ε, μια λέξη που λέγαμε ότι είχε εξαφανιστεί από το λεξιλόγιο, όμως το εξακολουθεί να σκοτώνει πολλούς ανθρώπους έβδομο αίτιο σε σημασία θνησιμότητα στον κόσμο είναι η φηματίωση. Τα τελευταία χρόνια δυστυχώς ο αριθμός των κρουσμάτων με φυματίωση που αντιστέκεται στα αντιβιωτικά αυξήθηκε. 9,4 εκατομμύρια νέα κρούσματα είχαμε στον κόσμο πέρσι. Κάθε δεύτερο άτομο έχει το βάκυλο του, ε, της φυματιώσεως στον κόσμο είναι στατιστικά στοιχεία, θα πρέπει να τα αναφέρουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, να καταλάβουμε καλύτερο ότι αυτή η ασθένεια σκοτώνει πάρα πολύ μεγάλο αριθμό Ευρωπαίων πολιτών. Κατάγουμε από μια χώρα που δυστυχώ είναι στη χειρότερη θέση όσον αφορά την ε, φυματίωση. Παρόλο τα τελευταία χρόνια υπήρξε μια μειωτική, ελαφρά μειωτική τάση, και μειώθηκε, μειώθηκαν τα κρούσματα φυματίωσης που αντιστέκεται στα φάρμακα, τα στοιχεία είναι άσχημα και εξακολουθούμε να ανησυχούμε. Χρειαζόμαστε συνεκτική σχεδιασμένη προσπάθεια για να ελεγχθεί αυτή η ασθένεια θα πρέπει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενώσεως να συνεχίσουμε τις δραστηριότητες που ασκήσαμε μέχρι τώρα, τους, ώστε να βελτιώσουμε τον έλεγχο της ασθένειας αυτής σε όλες τις χώρες, να βελτιωθεί η πρόσβαση στην περίθαλψη, στα φάρμακα, στην ποιότητα της μέρημνας τους ε, ασθενείς με φυματίωση. Θα πρέπει όλες οι κυβερνήσεις να καταλάβουν πόσο σημαντική αυτή είναι η μάχη και θα πρέπει να συνεργαστούμε του κοινωνικούς εταίρους όσο καλύτερα γίνεται η καταπολεμηθεί αυτή η ασθένεια που πιστεύαμε ότι ανήκε σε περασμένους αιώνε. Θα πρέπει να ε, κάνουμε τη μάχη, να δώσουμε τη μάχη μαζί σαν οικογένεια, να βοηθήσουμε ένα τον άλλον για να ξεπεράσουμε τη δυσκολία, διότι στο κάτω-κάτω είμαστε η Ευρωπαϊκή Ένωση και η δύναμή μα είναι στην ισχύ μα. Ευχαριστώ, Η κυρία το Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κανείς δεν θα πρέπει να πεθαίνει από τη φυματίωση. Έτσι είχε πει ο κ. Μπάνκι Μουν σήμερα ε, την ε, Διεθνή ημέρα της ε, καταπολέμησης ματιώσεως. Έχει δίκιο, αλλά πάρα πολύ, κυρίως οι φτωχοί και παιδιά στον κόσμο πεθαίνουν από τη φυματίωση. Γι' αυτό θα πρέπει να αυξήσουμε την υποστήριξη για το Διεθνές αυτό ταμείο που προσπαθεί να καταπολεμήσει την, την και την φυματίωση και την στον κόσμο. Όπως αναφέρθηκε, πεθαίνουν και άνθρωποι στην Ευρώπη από φυματίωση και θα πρέπει να πολεμήσουμε για να αποφύγουμε τη διάδοση, τη μετάδοση της φυματιώσεω που αντιστέκεται στα φάρμακα και να βρούμε αποτελεσματικό τρόπο να καταπολεμηθεί αυτή η ασθένεια ε, που αφορά όλους. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ε, Προστασία και Έλεγχο από τις Ασθένειες έχει σημαντικότατο ρόλο να διαδραματίσει και χαίρομαι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αναφερθεί σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, συνάδελφε. Συνάδελφε, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η πρόοδος της ιατρικής κάνει πολλά για να καταπολεμηθεί η φυματίωση. Κακώς θεωρούμε ότι είναι η ασθένεια των φτωχών χωρών. Γιατί στην Ευρώπη, στην Κεντρική και την Ανατολική υπάρχει σε ένα μεγάλο βαθμό και καμία χώρα δεν μπορεί να την αποφύγει. Εδώ και πολλές χιλιετίες. Πέρα από τους φάκελους που αντιστέχονται, πρέπει να φροντίσουμε να καταπολεμήσουμε την ασθένεια ολόκληρη. Πρώτα απ' όλα με την πρόληψη, με την παρακολούθηση στην ιατρική, με την έρευνα, με την εκλέκευση των μέτρων προστασίας, υγιεινής δηλαδή, συντονισμένα. Με δύο λόγια, πρέπει να στηριχτούμε στην καλύτερη δυνατόν στρατηγική. Όσον αφορά τη χρηματοδότηση τώρα μέτρων, πρέπει εδώ να κάνουμε μία διάκριση πρώτα απ' όλα στις χώρες μας, τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης πρέπει να είναι σε θέση να καλύψουν τα ιατρικά έξοδα. Όμως, στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι ασθενείς δεν είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τα έξοδα και χρειάζονται αλληλεγγύη. Από το 2002 λοιπόν έχουμε φροντίσει να την προσφέρουμε για τις ασθένειες αυτές, το AIDS, την ελονοσία και τη φυματίωση. Αν θέλουμε να μειώσουμε τις επιπτώσεις της φυματίωσης στο μισό από το 2000 μέχρι το 2015, πρέπει να δείξουμε αποφασιστικότητα υπέρ των ε, σεναρίων ε, που μας πρότεινε ο κύριος Κασίνσκι, ο πρόεδρος του Κέντρου Πρόληψης. Θέλω να ρωτήσω λοιπόν τον Επίτροπο προς ποια κατεύθυνση θα πάει, ποιο από τα τρία αυτά σενάρια προτείνει η Επιτροπή να ακολουθήσουμε για να καταπολεμηθεί η φυματίωση, η ελονοσία και το AIDS στο μέλλον. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Είναι δύσκολο να σας διακόψω μια που είναι τόσο αργά, αλλά πρέπει να το κάνω γιατί ε, πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμά μας. Η κυρία Καρβάλη έχει τώρα το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερόμαστε στην καταπολέμηση της σηματίωσης. Ήταν η μέρα αυτή σήμερα και είναι μια ευκαιρία να συζητήσουμε την εφαρμογή της σωστής πολιτικής και να συμμετάσχει η κοινωνία των πολιτών στη μάχη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ήθελε να μειωθεί ο αριθμός των κρουσμάτων της σηματίωσης. Στην Πορτογαλία όμως είναι πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα κρούσματα της φυματίωσης. Σήμερα που είναι η χρονιά καταπολεμήσεως της φυματιώσεως, σε κάποιες χώρες είδαμε να ξαναζωντανεύει αυτή η ασθένεια. Τα διάφορα σχέδια δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στρέφονται στην καταπολέμηση αυτής της ασθένειας. Θα θέλω να υπογραμμίσω τη σημασία που έχει η σχέση Ευρωπαϊκής Ενώσεως με τις αναπτυσσόμενες χώρες όσον αφορά τις κλινικές εξετάσεις και στα πλαίσια του προγράμματος πλαισίου για την ανάπτυξη ε, μέτρων κατά της Θα πρέπει να γίνει επιστημονική προσπάθεια και στις κλινικές έρευνες για την καταπολέμηση της φυματίωσης. Πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για να βελτιωθούν τα μέσα που έχουμε για την καταπολέμηση της φυματίωσης και για να προωθήσουμε νέες τεχνολογίες για τη διάγνωση για τα φάρμακα και για τα εμβόλια. Απευθύνω έκκληση λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις κυβερνήσεις να καταβάλουν τις δέουσες προσπάθειες για να δοθεί μεγαλύτερη μάχη κατά της ασθενείας για να μπορούμε επιτυχώς να την ελέγξουμε και να την εκριζώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί η φυματίωση, γιατί κάθε χρόνο περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι στον κόσμο πεθαίνουν και ένας στους τρεις στον κόσμο ε, είναι μολυσμένος με φυματίωση. Η φυματίωση είναι η πιο ευρέως διαδεδομένη μεταδοτική ασθένεια στον πλανήτη. Και αυτό σχετίζεται πολύ στενά με κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα αυτή η ασθένεια. Δηλαδή με τη φτώχεια, με την ανεργία, με τον αλκοολισμό, με το AIDS ε, με εξάρτηση από τα ναρκωτικά και με συστήματα στις, στις λιγότερα ανεπτυγμένες χώρες, συστήματα υγείας που δεν είναι καλά. Ε, θα πρέπει να εξαλειφθούν αυτοί οι παράγοντε που διευκολύνουν τη διάδοση τη ασθένεια. Τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, να θεσπίσουν κοινά μέτρα για την καταπολέμηση τη φρικτή αυτή ασθένεια. Θα πρέπει να υπάρξει κοινό πολιτικό διάλογο για οικονομική υποστήριξη και κοινό σχέδιο δράση. Θα ήθελα να πω ότι παρόλο που η φυματίωση συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των προτεραιατήτων για δράση, δεν χρηματοδοτείται επαρκώ η καταπολέμηση τη φυματίωσεω. Θα πρέπει να δοθούν τα αναγκαία ποσά και να προωθηθούν μέτρα για την καταπολέμηση ασθενεία. Συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της καταπολέμησης της φυματίωσης. Πρέπει να το θυμόμαστε. Εξακολουθεί να είναι πρόβλημα. Η φυματίωση, πάρα πολλοί άνθρωποι είναι μολυσμένοι με φυματίωση στον κόσμο και ε, από αυτούς από πάρα πολλοί ασθενούν βαριά. Θα πρέπει να υπάρχει σωστός έλεγχος Πρέπει να διαπιστώσουμε ότι παίζει σημαντικό η ρόλο κοινωνικο-οικονομική κατάσταση ευαλώτων ομάδων. Είναι κάτι, ένα στοιχείο που σχετίζεται με την ασθένεια. Θα πρέπει να υπάρχει σωστή περίθαλψη ελεγχόμενη περίθαλψη για την ασθένεια αυτή, ούτω ώστε να μειωθούν ε, τα διάφορα είδη της ασθένεια. Είναι πολύ δύσκολο βέβαια να βρεθούν και να τα κατάλληλα φάρμακα. Θα πρέπει τα συστήματα περίθαλψης να βελτιωθούν να παρακολουθούν τα κρούσματα κυρίως σε ευάλωτες ομάδες, να εκπαιδευτεί σωστά το προσωπικό πρόνοιας και θα πρέπει να διτεθούν και επαρκείς πόροι. 44 δις δολάρια θα πρέπει να τεθούν τα επόμενα χρόνια από το Ταμείο. Διαθέτουμε όμως τώρα, αυτό έχει προγραμματιστεί, τα μισά διαθέτουμε τώρα. Άρα, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με άλλου διεθνείς οργανισμούς για να πετύχει το στόχο και θα πρέπει να βοηθήσουμε τις χώρε του κόσμου. Ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στη διαδικασία του Κατσουδιάη. Δεν προσπαθεί κανένα να κινήσει το ενδιαφέρον μου. Λοιπόν, ο Επίτροπο Δάλη έχει το λόγο. Uh, Πρόεδρε, Έχοντας ακούσει τις παρεμβέσεις από τους ε, κυρίους βουλευτές, ε, θα ήθελα να σας ε, βεβαιώσω ότι η Κομισιόν λαμβάνει πάρα πολύ σοβαρά υπόψη το θέμα αυτό και λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη τις ιδέες που παρουσιάστηκαν εδώ στο Κοινοβούλιο μόλις τώρα. Είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε τους στόχους μας. Δηλαδή να θέσουμε υπό αυτή την ασθένεια. Αυτό το τύπο συζητήσεις είναι ιδιαίτερη σημασία για να μπορέσουμε να παραμείνουμε εστιασμένοι στην ασθένεια. Η συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και η υποστήριξη ημών είναι σημαντικότατη στις προσπάθειές μας για να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ασθένεια αυτή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες χώρες. Ευχαριστώ πολύ σε ευχαριστώ Επίτροπε κύριε Τελή. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση του θέματο. Το επόμενο σήμερα της ημερησιάτας είναι η παρουσία τη ακολούθηση του κυρίου Ένρικο Γερέδο Σαλόμ για τι επιπτώσει παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση σε αναπτυσσόμενε χώρε και την